τα οποία στηρίζει και η Επιτροπή Νομικών Θωμάτων αλλά και η Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία ε, Φράγα Εστέβεθ. Ε, ολοκληρώνεται η συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα. Ψηφοφορία λοιπόν αύριο στις 12. Αύριο Τετάρτη 6 Απριλίου συνεχίζεται η Ολομέλεια από τις 9 μέχρι τη 1, από τις 3 μέχρι τις 8. Θα σας μοιραστεί η μερίσια διάταξη, η οποία βρίσκεται και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού